Καλωσορίζω την Επιτροπή κυρία Κρούς και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η Ευρωπαϊκή, τα επόμενα βήματα. Η Χέλγα Τρούπελ είναι η συγκήτριά μας, έχει το λόγο. Χέλγα. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή θα έπρεπε να είναι το πολύ μεγάλο ψηφιακό σχέδιο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει Ευρωπαϊκά. Σημαίνει ε, μια ψηφιακή ε, βιβλιοθήκη η οποία ε, συμπεριλαμβάνει και ψηφιακά αρχεία. Όλα αυτά αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά και θα πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε ψηφιακά έργα όχι μόνο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τους πολίτες του κόσμου ολόκληρου. Η Ευρωπαϊκή έχει ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2008 ε, και χίλια ιδρύματα πολιτισμικά συνέβαλαν στην ίδρυσή της 180 εταιρικές οργανώσεις συμμετέχουν 6 εκατομμύρια έργων ευρωπαϊκών έχουν ψηφιοποιηθεί και πρέπει μέχρι το 2010 να φτάσουμε τα 10 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια μέχρι το 2015 ψηφιοποιημένων έργων. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο το οποίο είναι σημαντικότατο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι στιγμής από το πρόγραμμα ε, Content Plus και από τα κράτη-μέλη. Ε, οι συμβολές των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικές 40% για τη Γαλλία 16% για τη Γερμανία και πολλά άλλα κράτη-μέλη δίνουν πολύ μικρότερα ποσοστά ε, πρέπει πιστεύουμε να γίνει ε, το προπύργιο της ψηφιακής ευρωπαϊκής πολιτικής, της πολιτικής της Ένωσης δηλαδή. Πρόκειται για έναν πολιτισμικό δημόσιο θεσμό και για σαφέστατους λόγους θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει σωστός ανταγωνισμός με τα e-books, δηλαδή τα ψηφιακά βιβλία του Google γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει αμερικανικό μονοπόλιο, θα θέλουμε πραγματικά να έχουμε στην Ευρώπη την καλύτερη δυνατή προσφορά για την πολιτισμική μας ευρωπαϊκή κληρονομιά. Και επίσης θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας, ούτως ώστε οι πολίτες της Ευρώπης να μπορούν πραγματικά να έχουν μια επίδραση ε, σε αυτόν τον τομέα. Εφόσον πρόκειται για έργα εκτός δικαιωμάτων ε, πνευματικών, ε, πρόκειται για έργα δηλαδή κοινή κληρονομιάς, ε, τότε είναι διαφορετικό το θέμα, εντελώς διαφορετικό είναι όταν δεν υπάρχουν δικαιώματα και δεν προστατεύονται αυτά τα έργα Εάν θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαία να κάνει μια σωστή προσφορά για τα έργα τα οποία δεν δεσμεύονται από δικαιώματα δημιουργού θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα ε, τηλεχρησιμοποίησης αυτών των έργων για να υπάρχει ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά. Ε, ψηφιακή λοιπόν μορφή αποτελεσματική και ταχύτατη με διατήρηση ταυτοχρόνως των δικαιωμάτων του δημιουργού για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε συνενετικές λύσεις για όλα αυτά τα έργα που είναι πολύ ποικιλόμορφα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε στην περίπτωση ορφανών έργων τους έχοντες δικαιώματα. Ε, πρέπει να μιλήσουμε στη συνέχεια και για την στρατηγική του 2020 για μια εξέλιξη δηλαδή της κοινωνίας της γνώσης και της ψηφιακής κοινωνίας. Για, πρόκειται για την πολιτισμική ποικιλομορφία η οποία εξελίσσεται μέσα από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκά ε, που ε, ανήκει στο πρόγραμμα Ευρώπα 2020. Χρειάζεται μια κοινή πολιτική και κοινή κατεύθυνση. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από μια εκστρατεία για εξέβρεση χρηματοδότησης στον ιδιωτικό τομέα όπως υπάρχει και από το δημόσιο τομέα. Πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε ώστε οι πολίτες να μάθουν ότι υπάρχουν τέτοιες προσφορές. Πολλοί το αγνοούν και είναι ένα από τα έργα που πρέπει να αναλάβουμε η πληροφόρηση σχετικά. Στα πλαίσια του Catch the Eye, ο Πιότρ Μπόριτς είναι ο πρώτος μιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαίανα είναι ένα πραγματικό επίτευγμα που θα μας επιτρέψει να δώσουμε μεγαλύτερη ε, διάσταση στην ε, πολιτιστική μας κληρονομιά, να τη γνωρίσει περισσότερος κόσμος. Δεν πρόκειται για μια βιβλιοθήκη, αλλά για ένα ζωντανό μουσείο. ελπίζω να δημοσιευθούν και έργα όπως ας πούμε της Μαρίας ε, Κιουρί online. Αλλά προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς έργα χαμηλότερης ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε το copyright των ορφανών έργων και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες στα πλαίσια της ψηφιοποίησης ε, στα κράτη-μέλη, αν θέλουμε κάποια στιγμή να ταλαισφορήσει αυτό το πρόγραμμα. Ο κύριος Ενσίου είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ως εισηγητής ε, για την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΤΡΕ ε, για τα επόμενα βήματα θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την ε, πρωτοβουλία για την έκθεση και θα ήθελα να τονίσω ότι έχει συζητηθεί το θέμα και της δημιουργίας ιστοτόπων για βιβλιοθήκες, για, τη, για ψηφιακές βιβλιοθήκες, καθώς και για να προωθήσουμε ε, την διάχυση πληροφοριών μέσω των βιβλιοθηκών. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μία πλήρη έκθεση. Ελπίζω στο μέλλον η συζήτηση να συζητηθεί για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τους ιστοτόπους, την χρηματοδότηση και την οργάνωση ε, ενός μίας ε, ιστοπύλης. Θα ήθελα λοιπόν να μας απασχολήσει το θέμα για να δούμε τα ανωτέρω ζητήματα και να στεφθεί το όλο εγχείρημα από επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή θα μπορέσει να στεφθεί από επιτυχία πιστεύω και αποτελεί ένα κέντρο για πληροφορίες, πολιτισμικές πληροφορίες για την Ευρώπη. Ο κύριος Στάκουλα. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää oh, raportista. Muutenkin Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να συγχαρούμε την κυρία Τρούπελ για μια ε, εξαιρετική έκθεση. Πέρσι το θέμα αυτό συζητήθηκε από την Επιτροπή και νομίζω ότι το εγχείρημά της ήταν ε, εκπληκτικό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοια προγράμματα στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι μια κοινότητα αξιών. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε μια πολιτισμική κοινότητα. Έχουμε 27 μέλη με μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και νομίζω ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης πληροφοριών και έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Πιστεύω ότι ακόμα και οι μικροί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο έτσι ώστε να γνωστοποιήσουν την, τον πολιτισμό τους και έτσι ώστε να υπάρχει μια ισότητα για την προσβασιμότητα σε αυτά τα, τα δίκτυα. Moc dziękuję panie przedsedo. Moja grupa polityczna, ja osobiście e, nie jesteśmy specjalistami κύριε Πρόεδρε. Λέω ο κύριος Η πολιτική μου ομάδα και εγώ δεν είμαστε μεγάλοι υπέρμαχοι του πολλαπλασιασμού των γραφειοκρατικών προσπαθειών. Αλλά ευτυχώς για μας η Ευρωπαίανα, δεν είναι μια τέτοια προσπάθεια γραφειοκρατική. Ζούμε στην εποχή της εικόνας και όχι πια στην εποχή του γραπτού κειμένου και αυτή η κουλτούρα της εικόνας μας καθιστά χειρότερους πολίτες. Γιατί νομίζω μειώνει το επίπεδο της δημόσιας συζήτησης. Αν λοιπόν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, υπάρχει περίπτωση να μας κάνει καλύτερους πολίτες, νομίζω ότι τότε θα δημιουργήσει πραγματικά μια νέα γενιά καλύτερων πολιτών, οι οποίοι θα είναι πιο ενεργοί, πιο σοφοί και καλύτεροι άνθρωποι κιόλα. Ευχαριστώ κύριε Μιγκάλσκι. Ο κύριος Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παπα-Νικολάου. και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε για μια πρωτοβουλία που μπορεί να αποδειχθεί πραγματικός θησαυρό για την Ευρώπη. Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την εισηγήτρια, την κυρία Τρούπελ, για την εξαιρετική έκθεση που έχει υποβάλει. Αναφερόμαστε σε μια ηλεκτρονική πολιτιστική παρακαταθήκη των ευρωπαϊκών κρατών όπου θα επιτρέπει την πρόσβαση σε πρωτογενή πολιτιστικά στοιχεία. Και θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η επιτυχία της Europeana εξαρτάται από τη μορφή που τελικά θέλουμε να της προσδώσουμε. Και εννοώ ότι δεν θέλουμε μια Europeana αντίγραφο ηλεκτρονικών πλατφορμών που υφίστανται σήμερα όπω ε, ε, υπάρχει στο Google και το ε, ή το wikipedia. θέλουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πηγή τη οποία τα στοιχεία θα έχουν επιστημονική σημασία και χρησιμότητα μια πηγή όπου τα πνευματικά δικαιώματα θα προστατεύονται και η σοβαρότητα των περιεχομένων θα διασφαλίζεται. και αυτό νομίζω ότι με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και τη συζήτηση που έχουμε κάνει στην επιτροπή καλτ ε, εξασφαλίζεται. Εκείνο βεβαίω που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τελικά είναι το ενδιαφέρον των κρατών να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο για την προβολή του πολιτισμού του. Και εδώ οφείλουμε όλοι να αναπτύξουμε το ρόλο μα, να εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο στι εθνικέ μα κυβερνήσει, στου πολίτε των κρατών μελών, προκειμένου να ε, έχει απήχηση αυτό το έργο και να μπορούμε μεσοπρόθεσμα να το ε, αξιοποιούμε όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κυρίες και κύριοι, καταρχήν, για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Τρούπελ για αυτή την εξαιρετική έκθεση η οποία μας απασχολεί και συζητάμε. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόγραμμα έτσι ώστε ο ευρωπαϊκός ε, πολιτισμός να μπορέσει να ομαδοποιηθεί σε μια ψηφιακή ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε αυτό το όνειρο να στεφθεί από επιτυχία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει προσπελασιμότητα, γενικότερη προσπελασιμότητα σε αυτό, σε αυτό τον πολιτισμό. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα πολύ καλό ε, Συμβιβασμό για την Προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα έργα. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις προτάσεις που υποβάλλουμε και να τις ενσωματώσει στο δικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι για τη χώρα μου θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι αυτό που έχει σημασία είναι αυτά τα μεγάλα έργα να μην τα έχουμε σε τρεις βασικές γλώσσες, αλλά σε όλες. Όχι μόνο στα γαλλικά και στα γερμανικά, αλλά και στα πολωνικά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να μπορέσει αυτός ο πολιτισμός να μπει στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει κυρία Τικάου. Τα ωφέλη για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χάρη στην πρόσβαση στην Ευρωπαία είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό του ψηφιακού περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στις ευρωπαϊκές χώρες. Και επίσης και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο. Θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη μορφή αυτά τα έργα και πρόσβαση κατάλληλη για να αποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων με ειδικά προβλήματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά ασφάλειας των ιστοτόπων και διεκτυακών πυλών. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια βιώσιμη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος Ευρωπαίανα. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τα δικαιώματα των δημιουργών ε, έργων ψηφιακών. Ευχαριστώ και τώρα η Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη και δεν ξεχνώ και την κυρία Τρούπελ όλος ιδιαίτερος. Η έκθεσή σας μας έχει πραγματικά σαγηνεύσει. Είναι ευπρόσδεκτη. η ευρωπαίανα τα επόμενα βήματα ε, ξεκινάνε από ένα πολύ πλεονεκτικό σημείο αφετηρίας και υπάρχει και μια πολιτική στήριξη για την Ευρωπαίανα από πίσω. Καθώς αυτό αποτελεί το σημείο, ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης των ψηφιακών ε, έργων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τρούπελ, την εισηγήτρια, για τη δουλειά της θα ήθελα να τη συγχαρώ και για την ε, ονομασία που είναι μοναδική, Ευρωπαίανα. Ε, το όνομα μιλάει από μόνο του. Δεν χρειάζεται καν να το εξηγήσουμε. Η Κομισιόν ε, επίσης είναι και υπέρ του εναλλακτικού α, ψηφίσματος που έχει την ε, Συμφωνία των Βασικών Πολιτικών Ομάδων του Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι ε, αλλά είναι η αρχή, είναι η αφετηρία. Τα ψηφιακά βιβλία, χάρτες, ε, εφημερίδες, αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό και ηχητικά αρχεία ε, θα καταστούν προσπελάσιμα μέσω ίντερνετ από τον κόσμο. Και αυτό είναι βασικό για να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην, στον πολιτισμό σε μια ψηφιακή εποχή δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρθηκε από κάποιους ομιλητές, ε, από κάποιο ομιλητή ότι γινόμαστε καλύτεροι πολίτες. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Υπάρχει πάνω απ' όλα ε, η ευκαιρία να είμαστε πιο ευχαριστημένοι, να, ζήσουμε καλύτερα, να έχουμε μεγαλύτερη σχέση με την κουλτούρα, με τον πολιτισμό. Να ζήσουμε πιο ευχάριστα και πιο όμορφα. Και στην έκθεση της η Κομισιόν ε, τονίζει ότι είναι και ένα οικονομικό στοίχημα. Η ψηφιοποίηση και η online πρόσβαση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα δώσει πλεονεκτήματα σε διάφορες ε, δραστηριότητες, έρευνα, τουρισμό, εκπαίδευση και τα ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή είναι η συνιστόσα μιας ανευπροηγουμένου συνεργασίας ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων. Και όπως είπε σωστά η κυρία Τρούπελ, δίνει άμεση πρόσβαση σε 7 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα. Ας ξεκινήσουμε και ας προχωρήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η έκθεση του Κοινοβουλίου ε, τονίζει και διαφορετικούς τομείς προς τους οποίους θα πρέπει να κατευθυνθεί η Ευρωπαϊκή και αναφέρει και τις σχετικές πολιτικές όπου θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο ε, τα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη του, του ιστοτόπου εξαρτάται από την ε, συνεισφορά των κρατών μελών που θα πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να ψηφιοποιήσουν τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και να καταστήσουν όλα τα ψηφιακά αντικείμενα προσπελάσιμα μέσω του Ευρωπαίανα. Και χαίρομαι που το ε, Ευρωκοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν ενώνει τη φωνή του για να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κινηθούν πιο γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Το Κοινοβούλιο λέει ότι η Ευρωπαϊκή δεν θα πρέπει απλώς να δίνει πρόσβαση ε, σε έργα του δημόσιου χώρου, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και υλικό το οποίο προστατεύεται από copyright. Κυρία Τικάου, να σας απαντήσω. Πρέπει να βρούμε καλές λύσεις για να φέρουμε online έργα τα οποία έχουν εξαντληθεί. Να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ορφανών έργων, έργα τα οποία είναι αδύνατο να βρούμε τους συντάκτες, του, συντάκτες τους, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, η Ευρώπη κινδυνεύει σε λίγα χρόνια να μείνει πίσω, σε σύγκριση κυρίως με τις Ηνωμένες Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν κάνει μια μελέτη αντικτύπου για μια πιθανή νομική λύση για τα ορφανά έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συζητάμε τι θα μπορούσε να γίνει. Θα επανέλθω όμως αυτό όταν μιλήσω για την ψηφιακή ατζέντα. Γιατί είναι και ένα από τα θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Μια ενισχυμένη ε, εκδοχή του Ευρωπαίανα θα ξεκινήσει αργότερα με στη διάρκεια του χρόνου και θα δώσει πρόσβαση ε, σε πάνω από 10 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα. Το Κοινοβούλιο πολύ σωστά τονίζει ότι για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε τον ιστότοπο σε πολιτιστικούς φορείς ε, και σε κοινό. Οι πολιτικές δικηφορείς φυσικά ενδιαφέρονται όλος ιδιαίτερος γιατί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με τα έργα τους. Επίσης, να μην ξεχνάμε τους νεαρούς, τα παιδιά των σχολείων. Ε, είναι μια πολύ ευαίσθητη ομάδα και ενδιαφέρεται όλος ιδιαίτερος για το Ευρωπαίο. Θα πρέπει να ενδιαφέρεται. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντα θα εστιάσουμε πραγματικά ε, στην Ευρωπαϊκή. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα στη συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει στις Βρυξέλλες σε 15 μέρες στην ε, Ολομέλεια. Η επόμενη εισήγηση